υπάρχουν παρατηρήσει θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί μέσα διάταξη. Το πρώτο σημείο είναι η σύσταση δεύτερης ανάγνωσης του κυρίου Σικέρσκη για την διανομή τροφίμων σε άτομα χωρίς πόρους. Για τέσσερα λεπτά δίνω το λόγο στον κύριο Σικέρσκη. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Ε, κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα διανομής τροφίρων στους πλέον απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μακρά παράδοση. Το 1987 ξεκίνησε το πρόγραμμα όταν το Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει τα τρόφιμα διαθέσιμα στα κράτη-μέλη με την προϋπόθεση ότι θα διανέμονταν στους απόρους της εποχής εκείνης. Κατόπιν, τα επόμενα χρόνια, όταν τα αποθέματα τροφίμων είχαν αρχίσει να περιορίζονται, μπορούσε κανείς να αγοράσει αυτά τα προϊόντα από την αγορά. με την εξέλιξη της γεωργικής πολιτικής, τα αποθέματα παρέμβασης ε, περιορίζονταν διαρκώς, γι' αυτό χρειάστηκε να προβλέψουμε τη διάθεση περισσότερων τροφίμων στην αγορά. Η ε, απόφαση για την αγορά αναθεωρήθηκε, επανεξετάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που αποφάνθηκε ότι δεν συμβαδίζει με την νομική βάση που είχε προβλεφθεί και ότι το πρόγραμμα θα έπρεπε να περιορίζεται σε τρόφιμα που προέρχονται από τα αποθέματα παρέμβασης. Αυτό θα σήμαινε ότι από το 2012 και πέρα θα έπρεπε, θα είχαμε μόνο 100 ευρώ διαθέσιμα και όχι 100 εκατομμύρια και όχι 500 εκατομμύρια. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάστηκε να ενεργήσει. Στις 7 Ιουλίου πέρσι λοιπόν απευθύνθηκε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ζητώντας τους να προτείνουν μια λύση αποτελεσματική για τα επόμενα δύο χρόνια και να μην μειωθούν τα χρήματα τόσο πολύ. Πρέπει να θυμούμαστε ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής και η θέση του Κοινοβουλίου δεν είχαν γίνει δεκτές από το Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποφάσισε λοιπόν να προβλέψει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα συνέδε με την κοινωνική πολιτική αλλά το Συμβούλιο απέρριψε αυτό το σχέδιο πρότασης. Μόνο στη διάρκεια της πολωνικής προεδρίας ε, κατέστη δυνατή η αποδέσμευση του προγράμματος, του σχεδίου. Το Δεκέμβριο του 2011 έγινε ένα τριμερή διάλογο μεταξύ και, και Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δέχθηκαν την πρόταση του Συμβουλίου. Η Επιτροπή μας δέχθηκε τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου ως εκ τούτου στη διάρκεια μιας ολομέλειας στο Στρασβούργο. Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου ενέκρινε το σχέδιο κειμένου και όλα, το σύνολο επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια του Συμβουλίου που συνήλθε τον Ιανουάριο. Στις 26 Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο εξέφρασε την έγκρισή του στις προτάσεις του Συμβουλίου και συμφωνήσαμε να τα συζητήσουμε ε, τα θέματα αυτά στην Ολομέλεια. Η θέση αφορά το πρόγραμμα και πώς εφαρμόζεται φέτος και όπως θα εφαρμοστεί και του χρόνου τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Θα, ε, το ποσό των 500 εκατομμύρων ευρώ θα διατηρηθεί και μιλάμε για πολλά χρήματα. Η νομική βάση στα της ΚΑΠ, στηρίζεται στην ΚΑΠ και οι τροπολογίες μας, οι τροπολογίες που καταθέσαμε έγιναν δεκτές. Τα, ότι πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ε, τρόφιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε επίσης δεκτή και συμμετοχή της Ένωσης και υπάρχει υποχρέωση στα σημεία διανομής να αναφέρεται σαφώς η συμμετοχή της Ένωση της στο πρόγραμμα και η προέλευσή τους είναι κοινοτική. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να προστατεύσουμε, να βοηθήσουμε τους απόρους και τους ανέργους δεδομένων των ακραίων καιρικών συνθήκων που επικρατούν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στις στοχότερες χώρες χρειάζεται η παροχή βοήθειας. Υπάρχει ένας τεράστιος ρυθμός ατόμων μπορεί να ωφεληθεί από το πρόγραμμα, οι άστεγοι, τα ηλικιωμένα, τα υπερήλικα άτομα, αλλά και οι μονογονικές οικογένειες. Μετά από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αριθμός των απόρων αυξήθηκε 10 εκατομμύρια άτομα περίπου ζητού, ζουν κάτω από τη γραμμή της φτώχειας, το όριο της φτώχειας και άλλα 40 εκατομμύρια βρίσκονται σε κίνδυνο να ε, καταλήξουν στην ίδια κατάσταση. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις συμμετέχουν ενεργά στη προσπάθεια παροχής βοήθειας αυτών των ατόμων πρέπει να επιδείξουμε όλοι αλληλεγγύη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλέξουμε, επιλέξουμε την νομική βάση για την περίοδο 2014-2020. Ο Επίτροπος κ. Τσιόλος έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μία λύση μπόρεσε να εξευρεθεί για το έτη ε, 2012-2013 έτσι ώστε να συνεχίσει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Υπενθυμίζω πως πάνω από τρία χρόνια εντατικές ε, διαπραγματεύσεις ε, χρειάστηκαν και τελικά κατορθώσαμε να δώσουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο για αυτά τα προγράμματα για τα έτη 12-13 που δεν καλύπτονταν πλέον μετά από την απόφαση του δικαστηρίου. Φυσικά δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μία από τις σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας και δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν, ε, προσφεύγουν σε αυτά τα συστήματα αυξάνονται γεωμετρικώς. Ήταν, ήμασταν λοιπόν αναγκασμένοι και από ανθρωπιστικοπιάς να προσφέρουμε στους ε, άπορους. Ε, ευχαριστώ το Κοινοβούλιο το σύνολό του και ιδιαίτερα τα μέλη του Εργοκοινοβουλίου Κοινοβουλίου που ενεπλάκησαν υπέρ της συνέχισης ε, του προγράμματος. Επίσης, ε, χάρη στην δική σας στήριξη, ε, ένα συμβασμό σε αυτό το περίπλοκο ζήτημα μπόρεσε να εξευρεθεί χάρη δε στην έμονή σας και την ξεκάθαρη θέση που κρατήσατε. Να ευχαριστήσω επίσης με αυτήν την ευκαιρία και τα κράτη-μέλη που ε, δείχνοντας ευρωπαϊκό πνεύμα πραγματικά ε, εργάστηκαν για να πετύχουν ένα πολιτικό συμβασμό. Η Κομισιόν υποστηρίζει τα αποτελέσματα των διαθεσμικών διαπραγματεύσεων και ως εκ τούτου μπορεί να δεχτεί την θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση για να επιτρεπεί η συνέχιση του καθεστώτος μέχρι το 2013. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν δεν εφίστη κόπον για να καταστήσει δυνατή αυτή την ε, ε, εφαρμογή. Η πρώτη μας πρόταση το 2008 είχαμε προτείνει πολλές διορθώσεις ε, των κανονιστικών κειμένων για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και στις ενστάσεις ε, των κρατών μελών. Τώρα που υπάρχει η δική πλειοψηφία υπέρ της συνέχισης του προγράμματος για μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2013, τώρα λοιπόν υπάρχει η πολιτική συμφωνία και μετά την απόφαση, την κατάλληλη νομική βάση για να στοιχείψει το πρόγραμμα το 2012-2013 στο πλαίσιο της κοινή αγροτικής πολιτικής και να αποφύγουμε το πρόγραμμα να διακοπεί απότομα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να σας πω ότι οι υπηρεσίες μα θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα επιπλέον, επιπλέον πόροι για τα έτη 2012-2013 να δεσμευτούν το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα οι ομιλητές εξορμός των πολιτικών ομάδων για το ΕΛ και για δύο λεπτά η κυρία Λεπρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια συμφωνία επιτεύχθηκε λοιπόν και πρέπει, θα κληθούμε να αποφανθούμε αύριο στη διάρκεια αυτή της Ολομέλειας στο Στρασβούρο και πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά μου δημιουργούν μια περίεργη εντύπωση. Χαίρομαι βέβαια αρχικά, αλλά έχω και ερωτήματα και τέλος ανησυχώ. Χαίρομαι που οι Ευρωπαίοι που βρίσκονται σε ανέχεια φέτος και του χρόνου θα μπορέσουν να τραφούν χάρη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παροχής Βοήθειας στους Πόρους οι συμπολίτε μας δεν θα είχαν, ε, μπορούσαν να δεχθούν ότι τίποτε δεν γίνεται για να αποδεσμευθούν αυτά τα απαιτούμενα κονδύλια ενώ πληροφερηθήκαμε ότι 82 δισεκατομμύρια μη χρησιμο, παραμένουν χρησιμοποιητά στα ταμεία της Ένωσης. Διαρωτώ για το μέλλον του προγράμματος. Πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι από το 2014 θα διακοπεί η παροχή τροφίμων σε 13 περίπου εκατομμύρια απόρων Ευρωπαίων. Και πόσοι θα είναι τότε. Μπορεί ο αριθμός τους να έχει αυξηθεί σημαντικά. Υπάρχουν λύσεις. Τις γνωρίζουμε όλοι. Ας καλέσουμε λοιπόν το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του για να δώσει συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα στη διάρκεια του επόμενου πολιετούς πλαισίου διότι αν δεν συμβεί αυτό θα χρειαστεί να αναλάβουμε, θα δεχθούμε ε, μια θα υπάρξουν φοβερές συνέπειες. Ας υποστηρίξουμε λοιπόν όλοι μαζί τη συμβιβαστική λύση για τη διατήρηση του προγράμματος. Ευχαριστώ κυρία Λεμπρά. Από τη Σοσιαλιστική και Δημοκρατική Ομάδα για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Καπόλος Σάντσου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα φυσικά να υποστηρίξω τη σύσταση του συναδέλφου μας του κυρίου Σικέρσκ και να χαιρετήσω τον κύριο Τσόλος που εκπροσωπεί την Κομισιόν για την ε, αιμονή του να εξασφαλίσει την ε, βοήθεια αυτή προς τους πιο απόκληρους. Είναι απαραίτητο για τους Ευρωπαίους πολίτες να νιώσουν ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη η οποία τους αγκαλιάζει σε μια στιγμή ακριβώς που γίνεται όλο και πιο οξία η κρίση που διατρέχει την Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό το λόγο και παρά τις ε, αμφιβολίε ορισμένων κρατών μελών, εγώ είμαι πεπισμένο ότι θα μπορέσει να καταστηνατώ να διατηρηθεί αυτού του είδου η βοήθεια προς του φτωχότερου μέσα στον προπολογισμό. Δεν έχει σημασία αν θα είναι στον χώρο τη γεωργία ή σε άλλο κεφάλαιο. Το απαραίτητο είναι να διατηρηθεί και στο μέλλον αυτή η βοήθεια όσο υπάρχει φτώχεια στην Ευρώπη. Α ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα πάψει να υπάρχει αυτή η ένδια και θα έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε να έχουμε αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καπόλος για, τους δημοκρατι... για τη Δημοκρατική και Φιλελεύθερη Ομάδα. Δύο λεπτά κυρία Γκουλάρ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Έχω έρθει εδώ για την επίτευξη αυτού του καλού αποτελέσματος που είναι ένα καλό παράδειγμα ότι μπορεί να πετύχουν τα όργανα όταν συνεργάζονται και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη στα πλαίσια της διοργανικής διαπαραταξιακής ομάδας ε, της οποίας προεδρεύω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την επικουρικότητα και τι, ε, τι πάγεται σε κάθε επίπεδο απόφαση. Στην ομάδα μου υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ε, αντιμετωπίζουν την επικουρικότητα με πιο αυστηρό νομικό τρόπο ε, πρέπει όμως όλοι να φροντίσουμε τους απόρους και να μην αφήσουμε ε, την Ευρώπη να είναι μόνο το ε, θεσμικό όργανο που επιβάλλει προγράμματα λιτότητας χωρίς να παρέχει βοήθεια στις πιο ευάλωτες ομάδες της ε, κοινωνίας μας και ότι αυτό πρέπει να γίνεται μόνο σε το τοπικό και εθνικό επίπεδο. Με προβληματίζει το γεγονό ότι σαν πέρασματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την στρατηγική 2020 περάσαμε στο Europlus και δεν υπάρχει πλέον καμία αναφορά ε, ε, στον αποκλεισμό και στην ε, φτώχεια. Το θέμα της διατροφής πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής. Δεν έχω να προτείνω μια λύση, δεν λαμβάνω μια οριστική θέση σήμερα, αλλά υπάρχει και μια κοινωνική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη και κάτι που εξαρτάται από την κοινή αγροτική πολιτική κατά την άποψή μου. Του είδους διατροφής παρέχει η ΚΑΠ με σε τι κόστος σε εκείνους που δεν έχουν τα μέσα να αυτοχρηματοδοτηθούν. Πρέπει να στραφούν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις ή πρέπει να έχουμε μια ΚΑΠ που εξασφαλίζει διατροφή για όλους. Αυτό ήταν το πνεύμα των ιδρυτών της ΚΑΠ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά και υπολογίζουμε ότι θα μας βοηθήσετε κύριε Επίτροπε να έχουμε μια εκτεταμένη συζήτηση και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα για όλους. Ευχαριστώ κύριε Αγκουλάρ για τους πράσινους και την ε, ελεύθερη συμμαχία για ένα μισό λεπτό κύριος Χόουσλινγκ. Και εγώ θέλω να σας εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε καταλήξει με επιτυχία σε μια συμβαστική λύση. Είναι φανερό ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την παροχή τροφίμων στους φτωχούς και ιδίως σε μια στιγμή όπως τώρα που είναι περίπου 19 εκατομμύρια ατόμων τα οποία πλήττονται, τα οποία χρειάζονται μάλλον αυτή τη βοήθεια. Είναι μια απαραίτητη μορφή αλληλεγγύη από τη μεριά τη Ευρώπη. Θα πει, θα σκεφτούμε όμω θα σκεφτούμε και περισσότερο, όχι μονάχα για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά για την ανάπτυξη περαιτέρω προβλημάτων. Γιατί δεν είναι προφανέ ότι θα τελειώσει η κατάσταση αυτή φτώχεια. Και δεν θα είναι εύκολο να πούμε «Α, υπέρασε τώρα, δεν υπάρχει πρόβλημα». Δεν πρόκειται πια για μία ε, διάθεση ε, πλεονασμάτων αγροτικών όπως επρόκειτο στο παρελθόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα για μια εταιρική σχέση μεταξύ γεωργών και απόρων σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε τα άτομα αυτά τα οποία βρίσκονται σε συνθήκες ένδυας να μπορούν να βασίζονται σε αυτή την αρρωγή και επομένω να υπάρξει αυτή η εταιρική σχέση των γεωργών με τους ε, απόκληρους. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτή η μορφή τροφιμικής ε, βοήθειας να μπορέσει να έχει χρονική διάρκεια. Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι χώρες όπως η Γερμανία έχουν σταματήσει να προβάλλουν αντιρρήσεις. Ελπίζουμε θα μπορέσουν και αυτές να συνεργαστούν μέσα στα πλαίσια του νέου αυτού σχεδίου. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρος. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ένα λεπτό κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και εγώ δράτω με τις ευκαιρίες για να συγχαρώ τον κύριο Σιακέρσκι για την έκθεσή του. Πρέπει να πω όμως ότι αυτή η έκθεση ατενίζει προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Ανατρέχει στην εποχή που είχαμε βουνά βουτύρου και λίμνες γάλακτος κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώς έχει περάσει πια αυτή η εποχή, αν επιστρεπτεί. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε είναι μια κοινωνική πολιτική και δεν είναι πια ένα θέμα αγροτικής πολιτικής. Έχω απόλυτα, απόλυτη αλληλεγγύη με αυτούς οι οποίοι είναι άποροι και άστοιχοι αλλά πρέπει να υπάρξει και καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Το να αγοράζουμε τα τρόφιμα και τα διανέμουμε θα είναι πολύ ακριβό. Όπω είπα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ένα καλύτερο τρόπο και εδώ η Κομισιόν θα πρέπει να μελετήσει στο μέλλον ποια είναι η καλύτερη οδό. Και ξέρω ότι κάποιε χώρε έχουν προβλήματα οικονομικά αυτή τη στιγμή αλλά θα υπάρχουν πάντα άτομα τα οποία θα χρειάζονται βοήθεια. <coughs> επομένω. θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να δώσουμε την υποστήριξη. Ευχαριστώ κύριε Νίκολσον. Από την Ενωτική Αριστερά για 1,5 λεπτό ο κύριος Ομαρτζή, κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο μας ζητούν να ψηφίσουμε αύριο είναι η του 2014 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επιστήξης Βοήθειας στους Απόρους. Καμία εγγύηση δεν έχει χορηγηθεί μέχρι τούδε αναφορικά με τον μελλοντικό προγραμματισμό. Να το δηλώσουμε. Ντροπή. Μια ανασταλτική πλειοψηφία οργανώθηκε γύρω από την Γερμανία προκειμένου να παρεμποδίσει τους ποινώντε να τραφούν. Είναι λοιπόν ενδεικτικό στο ότι έχει συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θυσιάζει την αλληλεγγύη στο βωμό της ε, υπερφιλελεύθερης ε, πολιτικής και γραφειοκρατίας. Θα πρέπει να παραιτηθούμε να δεχτούμε μάλλον ότι το πρόγραμμα αυτό ε, δεν μπορεί να προχωρήσει με τις αποφάσεις που μου ληφθεί. Όταν όμως πρόκειται για κάποιες ε, φιλανθρωπίες ε, τότε ε, δημιουργούμε κάποια, κάποια εμπόδια νομικίστικα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω τα, οι θεσμοί μας έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Αυτή η απόφαση πραγματικά ε, επηρεάζει σημαντικά την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς σου. Ευχαριστώ κύριε ο Μαρτζή την Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας, ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα πέτυχε, αλλά δεν, στα, δεν σταμάτησε, γιατί η Κομισιόν τίποτα δεν σταματάει. Όχι μόνο αυτό, αλλά δρούν και παρανόμως. Το, η δανική Προεδρία είπε ότι αυτή η νομική βάση είναι εσφαλμένη. Γι' αυτό λοιπόν προτείνεται να τροποποιηθεί η κοινή αγροτική πολιτική, κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην μείωση των αγροτικών προϊόντων. Η Επιτροπή με κάνει να λυπάμαι για τους ε, Γάλλους ε, αγρότες. Στην ε, Ανατολική, στην East Anglia έχουμε πρόβλημα με την αγροτική παραγωγή. Η Κομισιόν λέει ότι οφείλεται στο το πρόβλημα του κλίματος και την θέρμανση του πλανήτη. Τελευταία άκουσα ότι δεν, έχουμε, δεν έχει ψηθεί η θερμοκρασία από το 2000 και μετά. Φέτος θυμάμαι τις χαμηλότερες θερμοκρασίες από το 1986 στην περιοχή μου. Οι προτάσεις της Κομισιόν είναι, ε, θα έλεγα, αφελείς θα, νομίζω θα πρέπει η κοινή λογική να υπερισχύσει. Mm. Ναι, ο κύριος... Ε, κοιτάξτε κύριε Άγνιου. Η λέξη stupid, αφελής, ίσως ε, να μην αρμόζει με την κοινοβουλευτική αυρότητα. Ο κύριος Στογιάννοβ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ ξεκινώντας ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάστηκε μόνο τέσσερις μήνες από την τελευταία κρόση να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο διαονιζόταν επί πολλά χρόνια σε επίπεδο Συμβουλίου. Αυτό που επιτεύθηκε είναι κάτι το θετικό και συμβαδίζει με το ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε. Αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας, διότι η περίοδος συμβιβασμού ε, έχει ξεπεράσει τα δύο χρόνια. Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα το πρόγραμμα, πρέπει αύριο να αρχίσουν προετοιμασίες για τη συνέχιση του στη διάρκεια της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας θυμίσω ότι η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα η οποία δεν έχει ακόμα συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχει μεν, ε, πληρώνει λεφτά, συνεισφέρει στο πρόγραμμα, αλλά δεν παίρνει τίποτε σε αντάλλαγμα. Εξασφαλίστε λοιπόν ότι όλες οι χώρες θα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Οι ομιλητέ τώρα, οι λοιποί ομιλητέ, καταρχήν για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Εράφ Γκαχία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πέραν των 80 εκατομμυρίων πτωχών για τους οποίους μιλάμε, είναι άλλα 43 εκατομμύρια ατόμων που έχουν δυσκολία για να έχουν πρόσβαση σε ζωικές πρωτεΐνες τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο γιατί αυτά τα άτομα μπορεί να μπουν <clears throat> στην ομάδα των ατόμων που βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της οικονομικής κρίσης. Επομένως είναι η κατάλληλη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα όχι με περικοπές στην επιστημιστική βοήθεια στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές η... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να υπάρξει <clears throat> μία περικοπή αυτής της βοήθειας, αλλά αυτό είναι και μια πράξη απόγνωσης μπροστά στην ε, αδράνεια και στην στάση εμπλοκής πολλών κρατών μελών τον τελευταίο καιρό. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν και πάλι πρωτοβουλίε ώστε από το 2014 να επανέλθει η επισητιστική αυτή βοήθεια. Δεν πρέπει να μείνουμε σταυρωμένα από τα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου για ένα τόσο σημαντικό θέμα από ανθρωπιστική έποψη. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να παραμείνουν έτσι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι διαπραγματεύσει για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικής σχεδίωσης για να τονίσουμε την απόψή μας και να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο Υπουργών που θα διατηρήσει τη βοήθεια αυτή προς τους φτωχότερους πέραν του 2014. Χάρη στην ευρωπαϊκή βοήθεια, οι τράπεζες τροφίμων έχουν κάνει ένα σημαντικό κοινωνικό έργο που δεν πρέπει να παραλύσει λόγω της ενέργειας ορισμένων ε, κυβερνήσεων. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες υπάρχουν εκατομμύρια ατόμων τα οποία έχουν κάπως καταφέρει να επιβιώσουν και έτσι δίνουμε και έμφαση στην ε, αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σάρμπου για ένα λεπτό. Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύση για αυτό το πρόγραμμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η φτώχεια αυξάνεται και εκατομμύρια άτομα δεν μπορούν πλέον να τρώνε ζεστή τροφή κάθε μέρα. 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ωφελήθηκαν από την επιστημική βοήθεια μέσω αυτού του προγράμματος και η μείωση των πόρων για τη χρηματοδότησή του ε, με βάση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς λόγω της οικονομικής κρίσης θα, ήταν, θα είχε καταστροφικές συνέπειες. Πρέπει να παραμείνει, να διατηρήσουμε αυτό το πρόγραμμα με χρηματοδότηση από την ΚΑΠ και μετά το 2013. Και θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ για τις γερμανικές και γαλλικές δηλώσεις σχετικά με την κατάργηση αυτού του προγράμματος. Η πρόσβαση σε είδη διατροφής είναι σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα, κυρίως σε περιόδους κρίσης. Πρέπει δε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους φτωχότερους πολίτες, να, τους να βοηθήσουμε τους ανήμπορους, που, που δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Αλληλεγγύη δεν είναι με όνομα αρχή που υπάρχει στο χαρτί. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Λάιον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, όπως δήλωσαν και συνάδελφοι σε αυτή τη συζήτηση, το πρόβλημα αυτό προκύπτει τη στιγμή όπου να βουτύρου και λίμνες γάλακτος ε, δεν ισχύουν πια. Και άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αλλαγή των συνθήκων και να αναγνωρίσουμε πως το πρόγραμμα αυτό ε, εμπίπτει στα πλαίσια της, κοινής, της κοινωνικής πολιτικής και όχι της αγροτικής. Η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να ε, αφορά την ε, κοινωνική πολιτική. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα αφορά τον επόμενο προπολογισμό για το προσεχές δηλαδή έτος ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιος συμβασμός. Αν δεν, μεταξύ των οργάνων, αν δεν υπάρχει αυτός ο συμβασμός, τότε τα, τα 500 εκατομμύρια θα μειωθούν σε 130 την επόμενη χρονιά, αφήνοντας 80.000 φτωχούς δίχως τη δυνατότητα να τύχουν στήριξη. Ειδικά σε αυτή την περίοδο κρίση το ζήτημα είναι κατεπήγον. Ζητώ από του συναδέλφου να στηρίξουν την προσωρινή αυτή λύση το πλαίσιο της αυριανής ψηφοφορίας. Αλλά αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τη συνέχιση του προγράμματος μετά το 2013. Αύριο θα ψηφίσουμε για μια μεταβατική λύση προκειμένου να απεμπλακεί η κατάσταση. Δεν είναι μια μακροπρόθεσμη λύση. Θα πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη, σωστή λύση για το πρόγραμμα αυτό και Επαναλαμβάνω το αίτημά μου δηλαδή να μεταφερθεί αυτό το πρόγραμμα στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Λάιον. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί αυτή η συμφωνία επιλύει ένα οξύ πρόβλημα. 18 εκατομμύρια Ευρωπαίων ιδιαίτερα πτωχών δεν θα είχαν καμία βοήθεια σε τρόφιμα χωρίς αυτή την απόφαση. Εξακολουθώ λοιπόν <clears throat> να ανησυχώ γιατί δεν υπάρχει ακόμα μια θετική προσέγγιση για το πώς θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις τράπεζες τροφίμων ώστε να απεξαρτηθούν από τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξακολουθεί να ελοχεύει ένας κίνδυνος. Κανείς δεν προετοιμάζει προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ότι μπορεί κάποτε αυτή η βοήθεια να μην συνεχίσει. Υπήρξε τώρα η παράταση του σχεδίου του μέτρου αυτού μέχρι το 2014, δύο χρόνια ακόμα. Αλλά το 2014 θα ξαναβρεθούμε σε αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που γνωρίσαμε τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Δηλαδή να είναι άδειε οι τράπεζε τροφίμων και να μην ξέρουμε πώ να ταΐσουμε του φτωχού. Αυτέ οι τράπεζε τροφίμων θα πρέπει να έχουν ίδιε δυνατότητα να συλλέγουν τρόφιμα τα αλλιώ, οποία αλλιώ θα πηγαίνανε στι χωματερέ. Είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια ανταλλαγή απόψεων με άλλου αυτόνομου οργανισμού, τράπεζε ε, τροφίμων, να υπάρχει επιμελητιακή βοήθεια και φορτηγά για τη μεταφορά των τροφίμων. Όλα αυτά απαιτούν μεγαλύτερη σαφήνεια, ιδίω για το χρονικό διάστημα επέκεινα του 2014. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν, το Συμβούλιο και οι συνάδελφοι να κινηθούν προ την κατεύθυνση αυτή. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Ταραμπέλα. Θέλετε να τη δεχτείτε βεβαίω, κύριε Ταραμπέλα. Θα ήθελα να πω τον κύριο Ταραμπέλα θα ήθελα να πω στον κύριο Λάιον ότι όταν ψηφίσουμε την ε, το six pack δεν θα είναι δυνατόν για τα κράτη-μέλη να έχουν μια κοινωνική πολιτική, διότι κάποιοι υπάλληλοι τη Επιτροπή δεν μπορούν να αυξήσουν τι κοινωνικέ δαπάνε εφόσον λειτουργούν μέσα από τον έλεγχο των δαπανών. Ρίχνουμε λοιπόν τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη που δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν μια κοινωνική πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν αυτό θέλατε να πείτε ή αν ότι πρέπει να ενεργήσουμε σε κοινωνικό επίπεδο και τον ευχαριστώ ήδη για την απάντησή του τον κύριο Λάιον. Μια διευκρίνηση για τον κύριο Ταραμπέλα. Θα ήθελα να είναι ευθύνη των κρατών μελών, αλλά δεν θα συμβεί αυτό. Γι' αυτό υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής, ώστε να γίνονται ορισμένα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μέσα με έχοντας οτομική βάση την κοινωνική πολιτική και όχι την αγροτική πολιτική. Για ένα λεπτό έχει το λόγο τους Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σουκένσκι για την εξαιρετική του έκθεση. Η επιστημιστική βοήθεια είναι πραγματικά απαραίτητη αφενός. Η φτώχεια ε, ε, απλώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φάνηκε φέτος. 600 άτομα πέθαναν, πέθαναν λόγω του ψύχους. Δεν υπάρχουν βεβαίω πλεονάσματα τροφίμων, αλλά ε, και υπάρχουν πλεονάσματα τροφίμων, αλλά, ε, αλλά η δυσκολία είναι στην ε, διάθεσή τους, στην εμπορία τους. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Η συνέχιση του προγράμματος το, μέχρι το 2014 είναι κάτι το σημαντικό και υποστηρίζω τον κύριο Νίκολσον και άλλους ομιλητές οι οποίοι είπαν ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να χρηματοδοτείται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και όχι στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής επειδή, επειδή οι στόχοι είναι διαφορετικοί Υπάρχει αφενός η παραγωγή τροφίμων και αφετέρου πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφα... επισητιστική ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί το πρόγραμμα και μετά αυτή την ε, διετή περίοδο. Για ένα λεπτό η κυρία Ζούμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία στοιχεία της ε, Eurostat δείχνουν ότι είναι δραματική κατάσταση ό,τι αφορά την ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 25% των παιδιών και 18% των ηλικιωμένων βρίσκονται σε κίνδυνο ένδυας. 115 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν το 24% του συνολικού πληθυσμού, απειλούνται από την ένδυα. Μετά από τον αντίκτυπο των λεγόμενων μέτρων λιτότητος θα υπάρξουν και περισσότερες επιπτώσεις με χαμηλότερες αποδοχές, μεγαλύτερη ανεργία, μείωση των κοινωνικών παροχών. Όλο αυτό το πλαίσιο επομένως είναι αποφασιστικό για να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η διανομή τροφίμων στα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ώστε να εγγυηθούμε ότι τα άτομα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να διατρέφονται και δεν θα θυγούν από την τροφιμική ένδια. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο μέσα στην επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020 να διατηρηθεί αυτή η επιδότηση τουλάχιστον στο τωρινό επίπεδο με την χρηματοδότηση 500 εκατομμύριων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση το χρόνο, τουλάχιστον. Ευχαριστώ κυρία Ζουμπέρ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Σκότας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε η σταθεροποίηση των τιμών και η στήριξη των πόρων είναι ένα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα αλλά και οι κρατικές αρχές έχουν υποστηρίξει αυτά τα προγράμματα μέσω διαφόρων προτάσεων, σηματοδότηση κλπ. Μιλήσετε και για ε, Σπατάλε στον τομέα των τροφίμων με τον κύριο Καρόνε εξετάσαμε το ζήτημα τη ε, ελληπού πρόσβασης ε, στα τρόφιμα από τους πλέον φτωχού. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Το να συμβάλλουμε στη μείωση των σπατάλη θα σημαίνει ότι βοηθάμε και τους πιο φτωχού τα άτομα που αντιμετωπίζουν ε, οικονομικές δυσκολίες ε, είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει λοιπόν ως εκ τούτου να βρεθεί χώρος ε, εντό των προγραμμάτων που μας απασχολούν. Θα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο, μια διοργάνωση με όσους μπορούν να βοηθήσουν. Θα ήθελα να ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή στην καθημερινότητα. Ευχαριστώ κύριε Σκότα. Το λόγο έχει για δύο λεπτά. Ο κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλησπέρα Επίτροπε. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο απέρα αυτού του επισητιστικού προγράμματος για τους ε, απόρους, αλλά έστω και αν αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, η συμβαστική αυτή λύση είναι ιδιαίτερα σπουδαία για αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Επί 25 χρόνια αυτό το πρόγραμμα έχει δείξει πόσο αποτελεσματικό είναι και πόσο πολύ βοήθησε τους απόρους. Πολλοί ωφελήθηκαν από την επιστημική βοήθεια στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να πω ότι Είμαστε το 400 κράτος στον κόσμο που υποφέρει από αυτές τις δυσκολίες με ανθρώπους που χρειάζονται επιστημιστική βοήθεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιδείξουμε συμπόνια και αλληλεγγύη και συγχαίρω τον εισηγητή για όλη τη δουλειά που έκανε, λέγοντα ταυτόχρονα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να, πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται για το μέλλον. Τι θα συμβεί μετά το 2013. Πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει την απαιτούμενη νομική βάση. Συμφωνώ με την Επιτροπή ω προ αυτό. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε ότι ένα στους τέσσερι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα στο μέλλον, στο παρελθόν η επιστημιστική βοήθεια στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, χρηματοδοτείται με 80 εκατομμύρια. Ένα στους 8 Αμερικανούς ωφελήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Μιλάμε λοιπόν για παραγωγικότητα, κοινοτομία και ανάπτυξη για το μέλλον και είμαι βέβαιο ότι αν βρούμε τις κατάλληλες λύσεις, τις σωστές λύσεις θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια. Πρέπει να παραμείνει για εκείνους που πραγματικά το χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νικουλέσκου για ένα λεπτό. Ο κύριος Ντεκάστρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη ικανοποίηση αύριο θα υπερψηφίσουμε την σύσταση για το δεύτερο πρόγραμμα διανομής ε, τρόφιμων τρεφούμεστων απόρων που λογοδέπει την παράτηση του χρόνου αυτού μέχρι το 2013. Μετά από όλους τους μήνες και με την εργασία πολλών και την δέσμευση αυτών θα τους ευχαριστήσω ξεκινώντας από τον Επίτροπο Σόλος και τον εισηγητή Σιχιέσκη. Κατορθώσαμε να πετύχουμε αυτό το σημαντικό ε, αποτέλεσμα που δεν εγκαταλείπει τους 18, 18 εκατομμύρια ε, φτωχών στην Ευρώπη. Η Πανελλημένη Κοινοβούλια αποφάνθηκε επί του προγράμματος και την παράτασή του μετά το 2013. Η πολιτική μας πρωτοβουλία ως εκ τούτου θα προχωρήσει. Εμείς δεν θα αρκεστούμε στην αυριανή υπερψήφιση, Πρόεδρε επόμενη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ευρώπη θα πρέπει να μπορέσει να συνεχίσει και στο μέλλον να είναι αλληλέγγυη με τους πλέον αδύναμους της κοινωνίας μας, ειδικά σε αυτή την περίοδο της σκληρής και επώδυνης οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ κύριε Κάστρο. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Αλουόρτ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, για την πίεση που έχει ασκήσει ώστε οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα βοηθήσουν άτομα <clears throat> τα οποία δεν καλύπτονται από την επιστημιστική βοήθεια το 2012-2013. Ζήτησε από την Κομισιόν πρόσφατα να δείξει, αν όχι συμπόνια, τουλάχιστον κοινή λογική για τη συνέχιση αυτού του σχεδίου. Χαίρομαι που θα συνεχιστεί για δύο χρόνια ακόμα, αλλά τα 13 εκατομμύρια άτομα που βασίζονται σε αυτό το πρόγραμμα θα χρειαστούν τη βοήθεια αυτή μετά από δύο χρόνια και μάλιστα οι αριθμοί του μάλλον θα αυξηθούν λόγω τη οικονομική κρίση. Πρέπει να υπάρχει μια τέτοια συνέχιση του προγράμματο, ώστε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση αλλιώ σε τρόφιμα θα μπορούν να καλύπτονται από αυτό το πρόβλημα. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα με θέματα επικορικότητα και επικάλυψη με εθνικού προπολογισμού, αλλά αυτό είναι ίσον μπροστά στον κίνδυνο τα άτομα αυτά να βρεθούν σε κατάσταση επιστηστική ένδυα. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν τι ιδεολογικέ ε, αντιπαραθέσεις. Τα 507 εκατομμύρια είναι πραγματικά πολύ σημαντικά για τα άτομα αυτά. Πρέπει να αφήσουμε στη, στην άκρη την πολιτική και τις πολιτικάτικες συμφωνίες και να σκεφτούμε αυτούς που δεν μπορούν να θρέψουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Για ένα λεπτό, η κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πάνω από 43 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απειλούνται ε, από τη φτώχεια και την έλλειψη τροφίμων. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε, ακούσαμε την παράταση του προγράμματος μέχρι το 2014. Οι φτωχότεροι θα εξακολουθούν να βρίσκουν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις την απαιτούμενη υποστήριξη που χρειάζονται καθώς οι ανάγκες θα αυξάνονται. Το σοβαρό το, το θέμα όμως είναι τι θα γίνει, τι θα συμβεί μετά το 2014. Η υπόσχεση ότι θα μειωθεί ε, η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το 2020 δεν είναι λέξη κενή. Πρέπει να βρούμε τους, τα μέσα και τους τρόπους να πετύχουμε αυτό το στόχο. Το νέο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να διονύσει το πρόβλημα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής ώστε τα κράτη-μέλη που έχουν ανάγκη να μπορούν να ωφεληθούν πραγματικά από αυτή τη βοήθεια. Αλλά υπάρχει μία προϋπόθεση. Αυτή η μεταφορά στο κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να συνοδευτεί με απαιτούμενο προπολογισμό για να μην εγκαταλειφθεί κανείς. Είναι θέμα αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Τέλος, κύριε Επίτροπε, οι φτωχότεροι δικαιούνται υγιή και ισορροπημένη διατροφή. Μόνο μία ΚΑΠ διάρκεια θα μα εξασφαλίσει ότι όλο και λιγότεροι Ευρωπαίοι θα χρειάζονται στο μέλλον την επιστημιστική βοήθεια. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο για ένα λεπτό έχει η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η διαθεσιμότητα τροφίμων για όλους τους πολίτες είναι κάτι το απαραίτητο για όλες τις ε, κοινωνίες, ε, τις πολιτισμένες. Αλλά εγώ αυτό το οποίο αμφιβάλλω είναι τα 500 εκατομμύρια κατά πόσον αρκούν για την απάντηση στα προβλήματα της ε, φτώχειας. Θεωρώ ότι αυτή την πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Η συνέχιση ενός προγράμματος ε, για τα επόμενα χρόνια δεν νομίζω ότι θα μας ε, γιάται πως θα είναι αποτελεσματικό. Με την συνέχιση λοιπόν αυτού του προγράμματος ε, σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης δεν βιώνουμε κατά πόσο θα βοηθήσουμε την ε, βιομηχανία παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου γιατί θα συμβεί εδώ. Ευχαριστώ κυρία Γκίρλινγκ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Σιμάνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όλο και περισσότερο άτομα, όλο και περισσότερα άτομα χρειάζονται επιστηστική βοήθεια. Και αυτό είναι απόρρια του χάσματος το οποίο διαβαίνεται συνέχεια μεταξύ φτωχών και πλουσίων στις κοινωνίες μας. Οι διαφορές υπάρχουν πάντα σε μια δημοκρατία, αλλά η, εν, η έντονη αυτή διαφορά μεταξύ φτωχών και πλουσίων σε μια κοινωνία δεν είναι κάτι το δικαιολογημένο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε την κατάλληλη μέθοδο για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτά τα οποία πράττονται σε εθνικό επίπεδο για να βοηθήσουν τους φτωχούς. Είναι συμπληρωματικό πρόγραμμα. Η αλληλεγγύη είναι μία από τις βασικές αρχές της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να περιορίσουμε την ένδια, αλλά δεν θα πρέπει να αυταπατώμεθα, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αποτελεσματικά και πλήρως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να απαρνηθεί αυτό το πρόγραμμα και, την κοινωνική, και στην κοινωνική της πολιτική. Πρέπει να θυμηθούμε όμως ότι πολλές οργανώσεις φιλανθρωπικές δεν περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν να τα πράξουν ό,τι μπορούν μόνες τους. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ. 18 εκατομμύρια Ευρωπαίων πλήττονται από την ένδια και εξατώνται από την επιστημιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι έτσι. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από τα πλεονάσματα της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής στο παρελθόν, όπως ανέφερε και ο εισηγητής ο κ. Σίκερσκι. Έχουν αλλάξει όμως οι καιροί. Έχουν πάψει να υπάρχουν αυτά τα αποθέματα. Η μεταβατική λύση που προτείνεται θα εξασφαλίσει την κατάσταση μόνο μέχρι το 2014. Το ερώτημα τι γίνεται μετά. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες. Δεν μπορεί η κοινή αγροτική πολιτική να παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες. Η κάθε χώρα έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις βασικές συνθήκες διαβίωσης για τους δικούς της πολίτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει, κύριε Ταραμπέλα, ότι αποκλείεται η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και τα εθνικά προγράμματα θα είναι βιώσιμα και θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Και αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Θα πρέπει, κύριε Επίτροπε, να κάνετε μια στρογγυλή τράπεζα με του εκπροσώπου των Εθνικών Κρατών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρείτε μια σωστή λυσιτελή στοχοθετημένη λύση για τα θέματα αυτά. Πρέπει επίσης να σταματήσουμε και τις, ε, τη σπατάλη των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ τα μισά καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Χρειαζόμαστε μια νέα κουλτούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε πληροφόρηση και σωστή αντιμετώπιση των τροφίμων. Το 1 τρίτο όλων των ενηλίκων δεν ξέρουν να μαγειρέψουν ένα αυγουλάκι. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι μια προϋπόθεση για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη διατροφή του πληθυσμού. Είναι ένα οικονομικό αλλά και κοινωνικό πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Κλάς. Για ένα λεπτό, ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Ο κύριος Ενέα έχει μια μπλε κάρτα. Κυρία Κλάς. Δέχεστε την μπλε κάρτα του κυρίου Ενέα. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Ε, το ότι πολλοί δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν τα τρόφιμα, αυτό σημαίνει ότι σπαταλούν και άρα αυτοί που δεν έχουν τίποτα δεν μπορούν να τραφούν. Λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να τραφεί, εξηγήστε μου, όταν έχουμε 0 ευρώ για να κάνουμε τα ψώνια μας. Κυρία Κλάς. Παρ' όλα αυτά είναι πιο λογικό και πιο ε, να τρέφεται κανείς με προϊόντα υγιή και βασικά. Και επομένω θα πρέπει να καταλάβει κανεί ότι με απλά πράγματα, με πατάτε, παραδείγματο χάρη, μπορεί να κάνει νόστιμα φαγητά. Έτσι είναι καλύτερο να αντιμετωπίσουμε την ένδια. Ε, Ευχαριστώ κυρία Κλάσ. Κύριε Ταραμπέλα, έχετε το λόγο τώρα. Δεν θα μιλήσω περί μαγειρικής, αλλά είμαι θλιμμένος σήμερα, θλιμμένος διότι έχουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτή δεν θα έρθει ποτέ να διεξαχθεί στη δύσκολη περίοδο που γνωρίζουμε σήμερα, διότι γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 500 εκατομμύρια ευρώ που ήδη βρίσκονται στον προπολογισμό, που θα μπορούσαν να αλλάξει ε, ε, να είχαν μεταφερθεί για να μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το καθήκον τους, δηλαδή να ανακουφίσει τα εκατομμύρια των ε, πολιτών μας, ε, που, των συμπολιτών μας που πεινούν. Και ο κύριος Μάρτς το είπε προλίγο. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια για τις τράπεζες και αρχίζουμε να τσιγκουνευόμαστε 500 εκατομμύρια για τους πιο φτωχούς. Είναι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Το μήνυμα που θα στείλει η Ευρώπη, αν διασώσουμε το πρόγραμμα για μετά το 2013, και σα συγχαίρω κύριε ε, ε, Επίτροπε, ε, για, να... για τη διάσωση μέχρι το 2013, αλλά από αύριο ξεκινάει ο αγώνα για να δούμε τι θα γίνει μετά το 2013. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψουμε το πρόβλημα αυτό που βοηθάει του ευτυχότερου πολίτε τη Ένωση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω ανάμεσά μας τον κύριο Πάξας. Δίνω το λόγο για ένα λεπτό στην κυρία Τόια. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πολύ θετικό το αποτέλεσμα που βρήκαμε για τη μεταβαρική περίοδο και εύχομαι να μπορέσουμε να βρούμε την οριστική λύση στις ε, δημοσιονομικές προοπτικές για μια απάντηση σταθερή, γρήγορη. Έχουμε ανάγκη από άμεση ενίσχυση διότι δυστυχώς ε, όλο και περισσότεροι φτωχοί δημιουργούνται στην Ευρώπη Σήμερα πολλοί δεν έχουν να τραφούν δεν, και δεν μπορούν να ζήσουν. Ε, ε, μιλάμε για μονογονικές οικογένειες, για χωρισμένα ζευγάρια λοιπά. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν του πολιτισμού ε, βλέπει το φάσμα της πείνας ενώπιόν της. Αυτό δεν θα πρέπει να μας καθησυχάζει όπως δεν θα μας όπως λένε κάποιοι συνάδελφοι, πρώτα θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες του τα κράτη-μέλη, να μάθουμε τον κόσμο να τρώει. Και μετά, εγώ λέω πρώτα θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την ε, ενίσχυση στους πιο άπορους διότι υπάρχει δυστυχώς μια Ευρώπη έξω από, τις, από τους χώρους αυτούς, αυτές και που ζητάνε μια Ευρώπη πιο δίκαια και πιο αλληλέγγυα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τόγια. Για ένα λεπτό ο κύριος Ταμπάτζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την μεγάλη χαρά οι φτωχοί και αυτοί οι οποίοι πεινάν δεν βρίσκονται σε αυτήν την συνεδρίαση γιατί θα νιώθανε πραγματικά ντροπή και αποστροφή προς τα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό πραγματικά είναι μια ντροπή και κάνω μια έκκληση για αυτούς που υποστηρίζουν το αγροτικό λόμπι. Και η Γεωργία δεν έχει καλό όνομα και καλή εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κύρος της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιωνόταν πάρα πολύ αν δεν θέλαμε εδώ πέρα <clears throat> να δώσουμε, να δώσουμε συνέχεια στη γεωργία σε βάρος του κοινωνικού τομέα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άμεσες πληρωμές του πρώτου πυλώνα περιλαμβάνουν ήδη πάρα πολλά κοινωνικά στοιχεία. Όποιος το αρνείται αυτό είναι ψεύτης. Γι' αυτό αυτοί οι οποίοι είναι φτωχοί και δεν έχουν <clears throat> να φάνε, δεν του νοιάζει καθόλου αν έρχεται το χρήμα από την κοινωνική πολιτική ή από την αγροτική πολιτική. Αυτό που του ενδιαφέρει να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και να φάνε. Γι' αυτό ζητώ από αυτού που υποστηρίζουν την γεωργική προσέγγιση να προστατεύσουν του φτωχού και τη γεωργία. Ευχαριστώ κύριε Ταμπατζή. Για ένα λεπτό. Η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμβατική λύση η οποία θα η έγκριση και η οποία θα μα επιτρέψει να συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό για δύο ακόμα χρόνια πριν από τι επόμενε πολιετέ δημοσιονομικέ προοπτικέ με το ίδιο επίπεδο υποστήριξη που θα δίνεται στου πιο φτωχού στην Ευρώπη. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ θα έρχονται 100% από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω ιδιαίτερα την ιδέα ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για προϊόντα εγχώρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για εισαγόμενες, εισαγόμενα προϊόντα. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε σταθερό αυτό το επίπεδο βοήθειας <clears throat> και ιδίως μέσα στην οικονομική κρίση, γιατί ο αριθμό των φτωχών έχει πράγματι αυξηθεί μέσα από την κρίση. Πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό μας, αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό στην τροφιμική βοήθεια. Είναι μεγάλος ο αριθμός των φτωχών και αυτών που έχουν ανάγκη τροφιμικής βοήθειας. Δεν έχει μειωθεί, έχει αυξηθεί μέσα στην κρίση. Αν εμείς μειώσουμε τη χρηματοδότηση, γυρίσουμε την πλάτη μας στους πολίτες μας και εγκαταλείπουμε τους στόχους να εξαλείψουμε την ένδια. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρεγέ πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι επιτέλου βρήκαν συμφωνία τα κράτη-μέλη που θα εξασφαλίσει τη συνέχιση του εψιστικού προγράμματος υπέρ των απόρων. Ήταν σημαντική αυτή η συμφωνία για τα εκατομμύρια Ευρωπαίων που μαθίζονται από την κρίση, αλλά δεν είναι ούτε κατά διάνοια ε, παρκέ. Τι θα γίνει μετά το 2014 σύμφωνα με την κυρία Μέρκελ δεν πρέπει πλέον να χρηματοδοτείται οποιαδήποτε κοινωνική παροχή και οποιοδήποτε κοινωνικό πρόγραμμα. Έχουμε κοινέ. Ε, ε, έχουμε ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα προστατεύσουμε. Η αξιοπρέπεια είναι το αντίθετο της ταπείνωσης. Κυρία Γκρελιέ, μήπως θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά για να σας προλαβαίνουν και οι διερμηνείς εννοώ, εννοώ πιο αργά, πιο αργά λέει ο πρόεδρος. Όχι πιο σιγά, πιο αργά. Διευκρινίζει. Η αξιοπρέπεια, έλεγα, είναι θεμελιώδη σκοπό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε αντίθεση με την ταπείνωση. Και το λέω αυτό στον ελληνικό λαό. Αξιοπρέπεια σημαίνει οι πολίτε να μπορούν να τρέφονται, να στεγάζονται και να ντύνονται αξιοπρεπώ, έστω πέρα από αυτά τα οποία λένε μικρά κράτη και κάποιε νομικέ δηλώσει. Καλό λοιπόν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βρουν λύση ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι στα πλαίσια τη Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ κυρία Γκρελή. Για ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Κάλενμπαχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Από τη μία πλευρά εγώ χαίρομαι που βρέθηκε μια λύση μεταβατική ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, την ε, τροφοδοσία των ενδεών με τρόφιμο μέχρι το 2014. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση πέρα από το 2013, από το 2014. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμπτωματική μονάχα πολιτική. Αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολεί είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η στάση ορισμένων πολιτικών ανδρών ή και γυναικών που οδηγεί πολλούς στη φτώχεια. Η φτώχεια και η ε, η έλλειψη πόρων στην Ευρώπη θα οδηγήσει σε μια καταστροφή στην Ευρώπη, όχι μόνο οικονομική και χρηματοπιστωτική καταστροφή. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ στην Ευρώπη μας αναγκάζουν να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζεται μονάχα να διανύμουμε τρόφιμα, να διανύμουμε και ευκαιρίες και να διανύμουμε και δικαιοσύνη, να δώσουμε ευκαιρίες για τους ανθρώπους να έχουν εργασία, να έχουν εισοδήματα. Όπως είπε και ο κύριος Καπόλεσσαμπ, ο στόχο είναι κάποτε να μην χρειάζονται πια αυτή τη βοήθεια. Να δώσουμε τώρα τρόφιμα για να αντιμετωπίσουμε την, την ένδια, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τι λύσει του προβλήματο ώστε να μην χρειάζονται τέτοια μέτρα στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέω ο Φτάνουμε στην οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία. 18 Οφθαλμοσυλλήπτε υπάρχουν. Και καταρχήν, σε πέντε θα δώσω το λόγο. προσπαθήσω να είμαι πιο ισορροπημένος. Θα δώσω σε εννέα οφθαλμοθυρευτές το λόγο. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Διάζε Μέρα. Θέλω να το ξαναπώ. Πρέπει να παρατεθεί το πρόγραμμα διαπάντα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε την αλληλεγγύη. Κανείς δεν θα μπορούσε να εξηγήσει μια αρνητική αντιμετώπιση. Γνωρίζουμε τα ποσά, τους αριθμούς αυτούς τους θλιβερούς. Τι σημασία έχει αν δίνεται από την ΚΑΠ ή από την κοινωνική πολιτική. Μπορούμε να εξηγήσουμε αυτό στους ε, συμπολίτες μας. Εγώ ούτε θέλω ούτε μπορώ. Πρέπει να δικαιολογήσουμε πώς τους αφαιρούμε αυτό που τους δίναμε μέχρι τώρα. Αυτό πραγματικά είναι ανεξήγητο. Ζητώ δικαιοσύνη και συμπόνια. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην δώσουμε αυτά τα 500 εκατομμύρια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και πλήττει τους πιο αδύναμους ε, γέρους, παιδιά, αστέγους, δίχως φάρμακα, δίχως τρόφιμα. Αντιδράστε κύριε του Συμβουλίου. Δεν βλέπω κανένα φτωχό στα έδρανα του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Ντιέρες Δεμέρα. Ο κύριος Δανέλης κύριε πρόεδρε η φτώχεια είναι ένα πολιτικό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. ασφαλώς η ευρώπη θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της φτώχειας. η ανακούφιση που δίνει το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους είναι σημαντική αλλά βεβαίως δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα και αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να καταργηθεί. επίσης τους απόρους δεν τους ενδιαφέρει εάν οι πόροι έρχονται από την καπ ή από το κοινωνικό ταμείο η τρέχουσα οικονομική κρίση στην ευρώπη θα επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης για μια νέα πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο βιώσιμο και συνεκτικό. η αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού είναι βέβαιο ότι είναι υπόθεση της ένωσης. παράλληλα θα πρέπει ίσως να θυμίσουμε ότι πρέπει να γίνουμε και πιο υπεύθυνοι ως πολίτες οι υπόλοιποι που έχουμε τη δυνατότητα να τρεφόμαστε επαρκώς τα 179 κιλά πεταμένης τροφής που αναλογούν στον κάθε πολίτη στον κάθε χρόνο νομίζω ότι αποτελούν ύβρι για τους απόρους και είναι ένα θέμα που πρέπει επίσης να μας απασχολεί. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δανέλη. Ο κύριος Μποβέ έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Μποβέ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σήμερα ορισμένοι δηλώνουν πως αυτό το πρόγραμμα δεν έχει τίποτα, ε, δεν έχει καμία σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική. Τους λέω όχι. Είναι σαφές ότι η κοινή αγροτική πολιτική που έχει ως στόχο την επιστημική ασφάλεια και τα προϊόντα να είναι προστά για το σύνολο των καναλωτών και ε, αφορά και το εισόδημα των γεωργών. Είναι λοιπόν ακρογωνίας λήθος της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής να τρέφει όλους τους πολίτες της. είμαστε ικανοί να μεταφέρουμε χρήματα για να, από την ΚΑΠ για να ε, χρηματοδοτούμε το ΙΤΕΡ ε, για 500 εκατομμύρια. Πώς ε, είναι δυνατόν λοιπόν να μην έχουμε δεν μην θέλουμε να διαθέσουμε 500 εκατομμύρια για την υποστήριξη των πλέον φτωχών. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να γίνει ένα συσχετισμό με σύνδεσμο ανάμεσα στην ΚΑΠ και την διατροφή των φτωχότερων. Θα πρέπει λοιπόν να δεσμευτούμε και ελπίζω ότι θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια πλαίσια τη κοινή αγροτική πολιτική ώστε και οι φτωχοί να έχουν πρόσβαση στην παραγωγή. Ευχαριστώ κύριε Μποδέ. Ο κύριο Ρούμπιξ. Ρούμπιξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εκατομμύρια φτωχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι για το γεγονός ότι η Κομισιόν μπόρεσε να βρει μια λύση με το Συμβούλιο για να παραταθεί το πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα παροχής τροφίμων στους φτωχούς. Είναι σημαντικό και για την ίδια τη γεωργία. Στη Λετωνία πέρσι υπήρξαν περίπου 185.000 άτομα τα οποία πήραν τέτοια επιστηστική βοήθεια. Ένα στου 12. Συμφωνώ με όλους αυτούς που λένε ότι πρέπει να παραταθεί αυτό το πρόγραμμα και να ισχύσει και στο μέλλον. και θέλω να εξασφαλίσουμε να έχουμε ε, τρόφιμα από τα αποθέματα παρέμβασης. Γιατί αυτά είναι τρόφιμα που ε, έχουν ήδη πληρωθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά πρέπει τα μέτρα αυτά να αφορούν μόνο τρόφιμα που παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, Επίτροπε, το Συμβούλιο σταμάτησε τη συνέχιση του προγράμματος ε, διανομής τροφίμων στους απόρους έρχισε η συζήτηση για το θέμα αυτό, ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα το 2012 και το 2013. Σαν προσωρινή λύση, οι αλλαγές που προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγιναν δεκτές η προμήθεια προϊόντων στα πλαίσια ανταγωνιστικών διαδικασιών, η προέλευση η ενωσιακή των τροφίμων. Δεν υπάρχει όμως λόγος να καθυστερεί το πρόγραμμα με νέες τροπολογίες. Πρέπει να τηρήσουμε την ετήσια οροφή των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική διανομή των τροφίμων, ώστε οι άποροι να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, Επίτροπε, πρέπει να αρχίσουμε δουλειά για το μηχανισμό που θα εφαρμοστεί στα πλαίσια του προγράμματος μετά το 2013, διότι αλλιώς οι άποροι δεν θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν αυτό το, το, ωφέλη αυτού του προγράμματος. Ευχαριστώ, κύριο Καλινόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια ζώνη ευημερία. Η οικονομική κρίση δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα, διαμαρτυρίες ε, και πολλοί ε, ζητούν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης ε, δείχνει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. 80 εκατομμύρια πολίτες την έχουν χρησιμοποιήσει. Δεν μιλάμε μόνο για μετανάστες, ε, αστέγους, ε, απόρους κλπ. 40 εκατομμύρια πολίτε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υποφέρουν από ένδια. Άλλοι τόσοι απειλούνται από αυτήν. Χαίρομαι λοιπόν που υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και θα μπορέσει επιτέλου να χορηγηθεί αυτή η βοήθεια δεν έχει σημασία η νομική βάση. Αυτό που έχει σημασία είναι η δέσμευση των θεσμών για τη βοήθεια που, που χορηγείται. Το λόγο έχει ο κυρίας Μουκόβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόσβαση στην τροφή θα πρέπει να είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα το οποίο θα γίνεται σεβαστό. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 2008 η βοήθεια χρησιμοποιήθηκε από 13 εκατομμύρια σε 18 κράτη-μέλη. Πάλι το 2010 ήδη είχαμε ανέβει σε 18 εκατομμύρια. Και η σημερινή κρίση οδηγεί σε περισσότερη ένδια τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το πρόγραμμα χρειάζεται να συνεχίσει να εφαρμόζεται και στο μέλλον για αυτούς που έχουν ανάγκη. Πάντως για το ένα παρόμοιο πρόγραμμα δεν πρέπει μόνο να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση αλλά να γίνεται και σωστή διανομή. Στην Σλοβακία μερικές φορές η διανομή καθυστερεί και αυτό ε, υπονομεύει το όλο πρόγραμμα. Όλη λοιπόν η αλυσίδα παροχής της βοήθειας θα πρέπει να οργανωθεί αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Κυρία Βολκόβα, κυρία Αντωνέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία. Πρόεδρε, κύριε... Κύριε Πίτροπε, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η τιμή των βασικών προϊόντων, τροφιμικού χαρακτήρα και αυτό σημαίνει ότι μειώθηκε και η αγοραστική δύναμη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κρίση είχε ένα πρόσθετο αρνητικό αποτέλεσμα. Αύξησε την, τρο τρωτή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φτωχότερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων είναι ένα θετικό μέτρο στο τωρινό πολιτικό πλαίσιο και μπορεί να δώσει μια σημαντική βοήθεια για 18 εκατομμύρια Ευρωπαίων χωρί να θίξει του ευθυνικού προπολογισμού. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν αυτή η μεταβατική λύση κατεπηγόντω μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό <clears throat> σχέδιο. Γιατί η πρόταση έχει ήδη μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Κομισιόν και τον Επίτροπο Τσόλος για όλες αυτές τις ε, προσπάθειες που κατέβαλα για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η βοήθεια και επίσης υποστηρίζω την πρόταση του ΕΛΚ σε σχέση με την παράταση του προγράμματος για να ενταθεί και σε επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ. Η τελευταία παρέμβαση είναι του κυρίου Όμπερ Μάιερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι καλό ότι υπάρχει αυτή η απόφαση να συνεχιστεί η βοήθεια. Δεν είναι μονάχα τα αποθέματα που θέλουμε να διαθέσουμε, γιατί αυτή η προβληματική έχει πάψει να υπάρχει. Ε, ο στόχος μας είναι φυσικά να μειώσουμε και το κόστος μεταφοράς τροφίμων το... και την επιβάρηση στο περιβάλλον. Θα ήταν πολύ καλύτερα να έχουμε τοπική παραγωγή και τοπική κατανάλωση προ... τροφίμων. Δεν θέλω να γυρίσουμε στα κολχώς και στα σοφχώς του κομμουνισμού, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια πιο οργανωμένη μορφή αντιμετώπισης της ένδυας, η οποία θα αυξήσει και τις θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα. Και δεν πιστεύει κανείς ότι θα μειωθεί τόσο γρήγορα η ένδυα, μάλλον θα έχουμε μεγαλύτερη φτώχεια στο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ κύριε Όμπερ Μάιερ. Ο κύριος Επίτροπος Τσιόλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εσύ, κύριοι κάποιες παρατηρήσεις μετά από τα σχόλιά σας. Το πρόγραμμα επιστημικής βοήθειας ε, στους άπορους ε, είναι ε, στόχος διπλό στόχο της κοινής αγροτικής πολιτική. Πρώτα απ' όλα, να διασφαλίσουμε ένα σταθερό και αξιοπρεπέ εισόδημα για του γεωργού, γι' αυτό έχουμε και τον μηχανισμό παρέμβαση, αλλά και από την άλλη πλευρά την δυνατότητα πρόσβαση όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρόφιμα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε. Αντί να καταστρέφουμε, έχουμε, δίνουμε την, παίρνουμε την παρέμβαση για να βοηθήσουμε του ε, πλέον ε, φτωχούς. Ε, φροντίζουμε να, φροντίζουμε να βελτιώσουμε και τα μέσα που έχουμε στο πλαίσιο κοινή αγροτική πολιτική. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν προτείνει διατήρηση του προγράμματο, διότι ακόμα και αν τα δημόσια αποθέματα δεν υπάρχουν, αλλά το ζήτημα τη πρόσβαση στην τρόφιμα δεν έχει ακόμα επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Κομισιόν προτείνει την συνέχιση του προγράμματος στο πλαίσιο της κοινωνικής ε, πολιτικής. Και δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, διότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σας το υπενθυμίζω. Δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν ε, ασκούν κοινωνική πολιτική. Αυτή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά αυτό δεν μας παρεμποδίσει να έχουμε κοινωνική πολιτική. Η απάντηση λοιπόν που δίνω σε όσους δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτό το πρόγραμμα μετά το 2014 Υπενθυμίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να διατηρηθεί ο προπολογισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Αυτή η πρόταση βρίσκεται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο που θα λάβουν απόφαση και σε συνάρτηση με αυτή την απόφαση η Κομισιόν φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν ε, απέρριψε ποτέ τις δυνατότητες που έχει για την ανάληψη πρωτοβουλίας ε, αυτό το πρόγραμμα για τους ε, απόρους ε, αφορά στην κοινωνική πολιτική αυτό δεν μας παρεμποδίζει να εξετάσουμε το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων, της διατροφής η Κομισιόν επίσης εξετάζει και τα ζητήματα αυτά και θα έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου με προτάσεις Καταλήγοντα, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Άγνιου που έκανε ένα σχόλιο προς την Κομισιόν. Σας διαβεβαιώνω κύριε Άγνιου ότι δεν ζήτησε ποτέ στους γεωργούς να παράγουν λιγότερο αλλά να παράγουν καλύτερα. Αυτό νομίζω ότι είναι ευφυές και όχι αφελές όπως είπατε. Ο κύριο Στογιάνοφ να πω ότι η Βουλγαρία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό είναι ε, απόφαση της κυβέρνησης της. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τις χώρες να συμμετέχουν, αλλά τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν μπορούν να το πράξουν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για την υποστήριξή σας ε, στο πρόγραμμα. Εκφράζω την ικανοποίησή μου ότι μπορούμε ήδη με αυτήν την απόφαση να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση του προγράμματος για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο ε, και το λόγο για να ολοκληρώσουμε το ζήτημα έχει ο κύριος Σικέρσκης, εγητής. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ήταν πολύ ωραίο να υπάρξει τόσο μεγάλη υποστήριξη υπέρ της συνέχισης αυτού του προγράμματος. Είμαστε νομίζω όλοι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικότερα για το γεγονός ότι ε, επέδειξε αποφασιστικότητα για τη διατήρηση του προγράμματος. Ε, ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νομική βάση ήταν αυτή που δημιούργησε πρόβλημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όχι η ιδέα του προγράμματος, η σύλληψη του προγράμματος, μόνο η νομική βάση αμφισβητήθηκε. Η νομική βάση δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τους απόρους, είναι γεγονός αυτό. Το Κοινοβούλιο ωστόσο πρέπει να αποφανθεί επ' αυτού και είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Μόνο οι χώρες που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτό, όπως μας είπε ο Επίτροπος. Η παρέμβαση είναι περιορισμένη αυτή τη στιγμή στις αγορές και προβλέπονται μεταρρυθμίσεις για το 2013 μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί για το πρόγραμμα μια νέα νομική βάση και είμαι πεπισμένος ότι θα βρει τη λύση το Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε επίσης, έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόζεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει να είναι εστιασμένο προς την επίτευξη αποτελεσμάτων Ίσως θα έπρεπε να έρθουμε σε επαφή με τις οργανώσεις διανομέων και με τις οργανώσεις καταναλωτών στις διάφορες χώρες για να μας πούν πώς θα μπορούσαμε να καταστήσουμε το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό. Πρέπει να συνεργαστούμε επίσης πιο στενά με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ας ευχηθούμε στους εαυτούς μας και σε όλες τις χώρες να μειωθεί όσο γίνεται ο αριθμός των απόρων. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία σε μια πρώτη φάση, διότι αυτό οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν και να τους παρακαλέσω να συνεχίσουν τις καλές τους προσπάθειες. Ευχαριστούμε κύριε Σιακέρσκη. ερχόμαστε στο επόμενο σημείο, η του κυρίου Νίκολσον